σύμφωνα με το κανονισμό 164 παράγραφο 2 δεν υπάρχει αίτημα να ψηφιστεί το χρονοδιάγραμμα. Θα περάσουμε τώρα στην, ε, στις ψηφοφορίες. Το επόμενο θέμα είναι η